της 15 Φεβρουαρίου. Προτείνω να εγκρίνουμε αυτές τις εντολές. Υπάρχουν παρατηρήσεις. Όχι, οπότε εγκρίνεται η κυριότητα αυτών των εντολών. Ο κύριος Ρότζερ Χέλμερ μου είπε πως δεν είναι πλέον μέλος της ομάδας ECR και από 5 Μαρτίου ανήκει στην ομάδα Ευρώπη για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία.